So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I think we Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ε, την ε, κανονική μας συνεδρίαση. Πρέπει να ξεκινήσουμε ε, να ψηφίζουμε. Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του Προέδρου θα ε, κάνω μια ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για οποιαδήποτε λάθη ενδεχομένως θα κάνω. Να μου πείτε αν κάτι δεν κάνω σωστά. Εάν κάτι δεν πάει καλά σίγουρα θα είναι δικό μου το λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, ε, μου ζητήθηκε αλλαγή ψηφοφορίας, μία ενιαία μοναδική ψηφοφορία σχετικά με το θέμα της συμφωνίας με τον Καναδά. Ε, είναι η εισηγητής ο Τσάρλ Τάνοκ, ε, είναι και η ισχυώδης εισηγήτρια υπέρ. Είναι το σημείο 20 το αρχικό της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Επιστρέφουμε τώρα στην ε, ε, έκθεση ε, σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία του 2016. Ο κύριος Φλέγκενστάιν θέλει να πει κάτι. Όχι. Ωραία. Επομένως, να ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ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 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 49 καταπίπτει. Τροπολογία 50 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά α, κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Να το το πρώτο λάθος. Εγκρίνεται, εγκρίνεται φυσικά. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 83, υπέρ, με την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, Άποχες. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 88 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε αν θέλετε. 149 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. <laughs> Προφανώς απορρίπτεται. 13 ψηφοί υπέρ, 47 κατά. Τρόπο, ε, συγγνώμη, συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 152 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της 152 Κόβατσεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 179. Άρχεται και πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 182 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω και εδώ ε, χρειάζεται επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την 182, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 30 ψήφι πέρα 31 κατά. Όπως και να έχει, θα είχε, ε, θα είχε καταψηφιστεί. Είμαστε τώρα στην 182, αυτή ψηφίζαμε, τώρα ψηφίζουμε την 186, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 187, υπέρ, κατά, αποχές. Και εδώ θα κάνουμε μια επαλήθευση για την τροπολογία 187. Άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 188. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι είναι σαφές ότι απερίφθη. Τροπολογία 191 υπέρ, κατά,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 κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές ε, 9 του κυρίου Κούκαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Α, έχει καταπέσει. Εντάξει, δεν το ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 13 του κυρίου Πιτίδιου. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 24 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Επαληθεύουμε λοιπόν την τροπολογία 26. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2 έχει αποσυρθεί. Υπαριθμών 3 μια εξαιρετική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε να περιθέσουμε την 4. Πολύ ωραία. 4 λοιπόν, τροπολογία 4. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται συγχαρητήρια Έντουαρτ. Η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έχουμε τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία της τροποποιημένης έκθεσης ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας και να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Κνούτ Φλεκενστάιν για την εξαίρετη έκθεσή του. to a... Λοιπόν, μια πολύ εύκολη χώρα ακολουθεί τώρα. Σχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Δεν ξέρω, εσύ θέλει να πει τίποτα, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χτες ευχαρίστησα όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιον που εργάζεται στη γραμματεία και θα φύγει ε, από τη γραμματεία ΑΦΕΤ. Ε, λέγεται Πέτερ Μπόιτοϊ και έχω συνεργαστεί μαζί του ε, στην έκθεση για την Ισλανδία 2009-2014 και μετά από το 2014 μέχρι σήμερα για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Είχαμε εξαιρετική αγαστή συνεργασία και καλή συνέχεια let's Πάμε λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το διεκπαιρεώσουμε γρήγορα. Με συμβαστική ένα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. η τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ τι είναι ονομαστική λέει Οι πράσινοι ζήτησαν ε, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Στην τροπολογία 2 τη συμβαστική είμαστε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθμών 80, το κύριο Σόλτες. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται έλεγχος. Ελέγχουμε την 80 παρακαλώ. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 90 του κυρίου Παπαδάκη. Κατά τμήματα είναι. Τμήμα πρώτον. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 102 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 5 υπέρ. 7 συγγνώμη κατά. αποχέ εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. αποχέ. Ελέγχουμε την 130 τώρα. Πέρας. Wow. Να σηκώνετε και κανένα χέρι για να σας βλέπω καλύτερα. Συμβαστική ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Παρακαλώ, απολυθεύουμε Εγκρίνεται. Τώρα. Γιατί την 143 έχουν ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλίση και αρχίζει τώρα. Ο κύριος Πρέντα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ονομαστική κλίση στη παρούσα διαδικασία. Ναι, το έχει ζητήσει πολιτική ομάδα για την 143. Α, καλά τότε. Ε, ας ψηφίσουμε τώρα. 143 ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη συμβαστική 10 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην τροπολογία 212. Ψηφί Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία σημαστική 18 Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 επε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 254 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 του κυρίου Τζαμπάσκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 288 κατά τμήματα. Οι πράσινοι έχουν ζητήσει αυτή τη χωριστή ψηφοφορία υπέρ της πρώτης κατά αποχές απορρίπτεται και οι πράσινοι ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα της 288 που αρχίζει τώρα. Ο εισηγητής λέει εγώ δεν έχω ιδέα για αυτά που λέτε τώρα. Δεν με είχαν ενημερώσει. Οι πράσινοι. Και τώρα τελειώνει η ψηφοφορία. Απερίφθη με μεγάλη διαφορά. Σαφέστατο. Ε, τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, δηλαδή εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος, 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 και 38 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θεέ μου, αναφωνεί ο πρόεδρος, oh my god. Λοιπόν, εντάξει, το διασκεδάζουμε κιόλας. Ε, έχουμε μια προφορική τροπολογία με ονομαστική κλίση που έχουν ζητήσει οι πράσινοι. Κύριε Σόλτες, διαδικαστικό είναι αυτό που θέλετε. Παρακαλώ. Πατήστε και κανένα κουμπάκι. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την προφορική τροπολογία. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την τροπολογία γενικώ. Επαναλαμβάνει ο κύριος Μπίχνερ, εμεί είμαστε ε, αντίθετοι με αυτή την προφορική τροπολογία. Να μην τεθεί λοιπόν σε ψήφιση. Ε, ωραία. Πάμε στη 40. Σόφκο. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μια στιγμή να δω τώρα τι γίνεται. Έχει ζητηθεί και άλλη ονομαστική ψηφοφορία από τους πρασίνους. Αγανάκτησε από τον εισηγητή. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια πράγματα, δεν με έχει ενημερώσει κανείς και είναι και περίεργα πράγματα. Ας ψηφίζουμε. Μα τι διαδικασία ακολουθούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ονομαστικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 40. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Απερίφθη 51-0. Well, perhaps somebody can explain... Μήπως μπορεί κανείς να μου εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Παρευρίσκεται η ομάδα των Πρασίνων. Ναι, εδώ είμαστε λένε. Λοιπόν, 41. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Στη 42. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα που πάμε. Στη 43. Ψηφί πέρα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 Αποχές. Απορρίπτεται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 και 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Wow. Φτάσαμε ήδη στην τροπολογία παρελθόν 4. Εγκρίθηκαν οι ένα και οι δύο, καταπίπτει η τρία. Καταπίπτει σας λέω και πάμε στην 4. Γι' αυτό ναι. καταχάρηκα. μπλοκ θέλετε. Ομού, όλες τις τροπολογίες αυτές. <laughs> Από την 4 μέχρι και την 9. Συμφωνείτε. Μέχρι και την 8, άντε. Είναι το μπλοκ Βιλίμσκι. Ψηφί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συλλήβδη. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 9. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Ωραία τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγχαρητήρια. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κατή μπλοκ τώρα, 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε πάλι το μπλοκ Βιλίμσκι από τη 16 μέχρι και την 22. Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Τι λέτε, τι θέλετε. Παρακαλώ, όχι. Όχι. Ωραία, μία-μία. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, φτάσαμε αισίω στην ε, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης, όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Συγχαρητήρια, κύριε Σεκητά. Εντυπωσιακή ψηφοφορία. So, bravo. Συνεχίζουμε. Τι κάνουμε τώρα. Why don't you give me yours? Next vote, we come. Επόμενη έκθεση. Σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή του 2015 για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εισηγητή τον κύριο Μπαλτσίτη. Θέλετε να πείτε τίποτα? Δεν είστε εδώ. Εντάξει. Ξεκινάμε. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δύο έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 7, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε. 9. πέρας εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, Εποχέ. Ε, απορρίπτεται. 13, 12 υπέρ, κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, Εποχέ. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Και 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. Επόμενη. Περνάμε τώρα στην απαλλαγή Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για το δημοσιονομικό έτο 2015. Είναι το τμήμα 10. Ο εισηγητή δεν είναι εδώ, ψηφίζουμε. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 5 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα, επόμενη έκθεση. Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των Καταμαλών τη αφενό και τη Δημοκρατία του Λιβάνου αφετέρου για να ληφθεί υπόψη προσχώρηση τη Δημοκρατία του Κρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια, κυρία Μανέσκου. Θέλετε να πείτε τίποτα, συγγήτρια. Ωραία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη. Αυτό ήτανε. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες για σήμερα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό το εγχείρημα. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγο πιο μπροστά από το πρόγραμμά μας, οπότε θα περάσουμε τώρα στο σημείο 21, ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη της αντοχώκ αντιπροσωπείας της ΑΦΕΤ στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και την Ιορδανία. 2 έως 6 Ιανουαρίου. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Η αποστολή αυτή ξεκίνησε, έγινε μάλλον στις αρχές της χρονιάς. Προείδρευσε ο κύριος Μπροκ. Και ήμουν και εγώ εκεί, ήμουν μέλο αυτή τη ad hoc αντιπροσωπεία. Είχαμε πολύ καλέ και επικοδομητικέ συζητήσει στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, στα κατεχόμενα. στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η αντιπροσωπεία ταξίδευσε στην Παλαιστίνη και θα δώσω στους συμμετέχοντες αντιπροσωπείας το λόγο και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπρόκ τον ίδιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιτ. Είναι παρόντε σχεδόν όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας. Οπότε δεν θέλω να σας κουράσω. Θα είμαι σύντομο, όπως είπες πήγαμε στην Ιερουσαλήμ στη Ραμάλα και στο Αμάν για μία μέρα κάθε φορά. Εκεί ε, κυριάρχησαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα σεμινάριο στη Γνεσέτ με τους συναδέλφους της Ισραηλινής Βουλής Κυρίως πρόκειται εκεί για το ρόλο του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας στους πολέμους δι' αντιπροσώπων, το θέμα ε, των ε, ξένων μαχητών και ο επικίνδυνος ρόλος ε, στη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά που προκαλεί εκεί η Χαμάς. Και συμφωνήσαμε όλοι ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και προς τους δύο, και προς το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Ε, αγαπητοί Κροάτες συνάδελφοι, δεν θέλω να σας ενοχλήσω εκεί στο κροατικό λόμπι, αλλά μήπως θα θέλατε να συνεχίσετε έξω τις ε, συζητήσεις σας. Κύριε Μπρόκ, παρακαλώ συνεχίστε. Τώρα φύγαν και οι τελευταίοι κρότε. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία ότι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τους πόλεμους, πολέμους συγγνώμη, αντιπροσώπων που ε, διεξάγουν στην Ιεμένη, στο Ιράκ και στη Συρία το Ισραήλ θεωρεί ότι υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή από το Ιράν προς τη Σιητική κυβέρνηση του Ιράκ να συνεργάζεται και με τον Άσαντ και με τη Χεσμολάχ, ότι υπάρχει μια ενιαία γραμμή, αυτά λέει ε, ο, ε, Ισραηλινή γραμμή και ε, ε, αυτοί οι Σιήτες συνεργάζονται λέει και με τη Ρωσία. Και στην ευτική διαδικασία στη Συρία και στο Ιράκ η Δύση μάλλον δεν έχει προτείνει πρωταγωνιστικό ρόλο και προσπαθούν κάποιοι de facto να παρουσιάσουν ε, την ε, Ρωσία ως το μόνο ειρηνοποιό εκεί στην περιοχή. Βλέπε και τη συνάντηση στο Καζαχστάν που επρόκειτο να, μετα... επακολουθήσει ε, μετά από την επίσκεψή μας με πρακτική απουσία των Ευρωπαίων και ανησυχεί το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά μας είπανε στη Ραμάλα και το καταλάβαμε και από το ίδιο το Μεσανατολικό, από τις διάφορες συναντήσεις, συναντιόνται και ε, κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι δεν θέλει τις συναντήσεις. Και η διαμεσολάβηση γίνεται κυρίως μέσω της Μόσχας. Δεν ξεπλάγει πόσες φορές έχουν πάει οι Ισραηλινοί στη Μόσχα. Και πάλι βλέπουμε ότι στην παγκόσμια στρατηγική έχουμε κάπου ισορροπίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, πρωταγωνιστεί σε τέτοιες συνευτικές διαδικασίες, στην άμεση γειτονία μας, έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στο Ισραήλ η συζήτηση και για αυτό το θέμα και για άλλα διαφέρει ε, ανάλογα με το αν στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Στον Ισραήλ τουλάχιστον περίμεναν τότε με μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Ο υπουργό ε, Δικαιοσύνης Μπένετ ε, που εκπροσωπεί τους ε, τον χαρακτήρισε έτσι και ο, Πρωθυπουργός Νετανιάχου και μίλησε για τη μεταφορά ε, της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ ε, στην Ιερουσαλήμ. Και μόλις βγήκε ο Τραμπ, αποφάσισε το Ισραήλ να επεκτείνει τους οικισμούς των επίκων και ασκήθηκε τεράστια κριτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για το ψήφισμα του ΟΗΕ, ότι είχαν ε, ε, εκφράσει επικρίσεις για τους επικισμούς. Ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν βάλει βέτο. Στη Δυτική Όχθη τώρα, πήγαμε στην ε, περιοχή City λεγόμενη γύρω από τη Βιθλεέμ, όπου είναι δήμαρχος μια χριστιανή Παλαιστίνια. Στο μεταξύ η Βιθλεέμ δεν απομονώνεται από την Ιερουσαλήμ μόνο με το τείχος που έχει σηκώσει το ε, Ισραήλ, αλλά την έχουν και περικυκλώσει γύρω-γύρω την πόλη για να μην μπορεί να επικοινωνεί με την περιοχή C, area που ε, έχουν αναπτυχθεί οι οικισμοί. Και πραγματικά αυτή η περιοχή C είναι το 60% της δυτικής όχθης. Μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για παλαιστινιακό κράτος από πλευράς εδαφικής και μόνο. Η κυβέρνηση στη Ραμάλα δεν έχει την παραμικρή επιρροή του έλεγχο καθόλου στη ζώνη εκεί. Με άλλα λόγια τι σημαίνει αυτό. Ότι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στο μεταξύ όπου η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ελέγχει ούτε τη Γάζα, γιατί εκεί την ελέγχει η Χαμάς, έχουμε μια κατάσταση που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μεγάλα τμήματα ε, της δυτικής όχθης να ελεγχθούν, γιατί αλλάζει και η δημογραφία με την πολιτική του επικισμού και σιγά σιγά ε, αρχίζουν να χάνουν την πίστη τους ε, στην ίδια την δυνατότητα να υπάρχει κράτος δεν είναι μόνο η βούληση που δεν υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται και επικράτεια πια για κράτο. Και όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να το δεχτούν. Εμεί είμαστε υπέρ τη λύση δύο κρατών, όπω κατά τα άλλα και η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Με όσου συζήτησα, δημερώ είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο και τους προέδρους ε, κομμάτων της αντιπολίτευση και έχουν αντίστοιχη τεράστια ανησυχία για το κατά πόσο ε, δεν υπάρχει καν συζήτηση για τα δύο κράτη, όχι μόνο ως πραγματικότητα, αλλά και ως υπόθεση. Και θα υπάρξουν μεγάλες συγκρούσεις νέες ή ιστοδυνικές. Ο δημογραφικός παράγων και μόνο θα οδηγήσει στο να είναι μειονότητα Ισραηλινή στο ίδιο του κράτος ή θα φροντίσει να δημιουργηθεί ένα apartheid γιατί αν η πλειοψηφία, η πλειονότητα του λαού σε μια χώρα, ε, του πληθυσμού δεν έχει δικαίωμα ψήφου, τότε αυτό μπορεί να έχει συνέπειες. Λοιπόν, περιγράφω την κατάσταση όπως την είδαμε εκεί και τη συμμερίζονται και πολλοί άλλοι. Οπότε, πραγματικά στη Ραμάλα είδαμε απελπισία και απόγνωση. Ε, και ματέωση, που μπορεί να μην είναι η καλύτερη των ανθρώπων, αλλά είναι πιο μετριοπαθής από τη Χαμάς και σε 20 χρόνια δεν έχουν καταφέρει τίποτα οι πιο μετριοπαθείς. Ε, στην Ιορδανία ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψής μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε με τον ε, ε, ε τη βασιλέα, γιατί ο βασιλιάς ήταν ε, διακοπές με τον πρίγκιπα Φαϊσάλ. Ε, ο αντιβασιλέας ε, προέρχεται από το στρατό, μας εξήγησε τα θέματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και μας είπε ότι λόγω της πίεσης του ίσης στην Ιρά, Ιράκ και στη Συρία, αν προχωρήσει προς τον Νότο θα μπει και στην Ιορδανία. Και όλο και περισσότερο αυξάνονται οι πρόσφυγες σε μια χώρα που είναι πάρα υπάρχει μια περιοχή στα σύνορα ε, ε, Συρίας-Ιορδανίας όπου δεν μπορεί να περάσει κανένας πρόσφυγας πια και μας λένε ότι ανησυχούν για τη σταθερότητά τους και αν τερματιστεί και η λύση των δύο κρατών από τη μια και από την άλλη επέλθει μια κατάσταση όπου μεταφερθεί και η πρεσβεία μας λένε εμείς πώς θα το συγκρατήσουμε αυτό δηλαδή ακούμε φωνές από την Ιορδανία ότι ανησυχούν Μήπω υπάρξει ρίζοσπαστικοποίηση και στην Ιορδανία την ίδια. Αν κοιτάξετε το χάρτη, αυτά είναι πάρα πολύ σκούρα πράγματα γιατί όλες αυτές τις δεκαετίες ε, ήταν η θέση της Ιορδανίας πάντα συγκρατημένη, λογική. Αν πιεστεί το καθεστώς εκεί μπορεί να υπάρξει αστάθεια και προβλήματα που δεν έχουμε ενδεχομένως ακόμα διανοηθεί. Και θα πρέπει να φροντίσουμε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει με προγράμματα έτσι ώστε να ε, αφαιρεθεί κάποια πίεση από την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στην Ιορδανία για να αποσοβηθούν τέτοιες καταστάσεις που μπορεί να είναι λόγω της φτώχειας, λόγω της λειψιδρίας, λόγω της τρομοκρατίας, λόγω του προσφυγικού, υφίστανται τεράστιες πιέσεις. Και μπορούν τα πράγματα να εκτροχιαστούν. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Φεύγοντας από εκεί, δεν γύρισα αισιόδοξο πάντως και γεμάτος ελπίδες. Δεν ξέρω άλλοι συνάδελφοι αν το βλέπουν διαφορετικά. που μπορεί να είναι πιο αισιόδοξοι και να βλέπουν καλύτερα το μέλλον ε, από μένα, με μεγαλύτερη ενόραση. Ευχαριστώ πολύ, Αλμαρ Μπρόκ. Ε, ήθελα να ζητήσω από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην Ανθόκα προσωπία, να μας πούν τις εντυπώσεις τους. Ποιος θέλει το λόγο. Έχουμε αρκετούς ομιλητές. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Έλμαρ Μπρόκ ήδη ανέφερε τα σημεία τα οποία ήταν τα πλέον σημαντικά, τις επαφές που είχαμε επί τόπου. Πρέπει να πω ότι στις τρεις μέρες ε, ε, είχαμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ εντατικό, είχαμε πολλές συναντήσεις και αντιπροσωπείς κτλ. Και να σας πω τώρα κάποια στοιχεία τα οποία θεώρησα σημαντικά. Πρώτα απ' όλα το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο ετέθη ε, και από τους συνομιλητές αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα στην Ισραήλ και στο Αμάν. Όταν οι φίλοι Ισραηλοί αναφέρονται σε τρομοκρατία, ε, η πρώτη τους ε, αναφορά είναι οι Σιήτες, ε, το Χεσμπολά, αυτοί είναι οι τρομοκράτες για τους Ισραηλινούς. Όταν όμως φτάσει κανείς στο Αμάν, οι φόβοι αλλάζουν. Φοβούνται τους Σουνίτες που ίσως θα ασκήσουν πιέσεις στα σύνορα εάν σημαντικές πόλεις όπως ε, η Ράκα πούμε ε, πέσουν και επομένως ε, υπάρξουν κύματα προσφύγων αλλά και τρομοκρατών που θα περάσουν στο Ιορδανικό έδαφος γιατί το πρόβλημα των συνόρων είναι μεγάλο για την Ιορδανία. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο ετέθη ε, και στο Αμάν και στη Ραμάλα και παντού αυτή η νέα σχέση ανάμεσα σε Ιρανούς, Τούρκους ε, και ε, Ρώσους όσον αφορά τη διαχείριση του Συριακού προβλήματος και τον ε, φόβο που εκφράστηκε, με διαφορετικό τρόπο βέβαια κάθε φορά, ε, όσον αφορά ε, μια επίλυση ενδεχόμενη του προβλήματος χωρίς συμμετοχή των Αράβων. Και ακούσαμε διάφορα σενάρια όσον αφορά αυτό το ζήτημα συμπεριλαμβανομένου, συμπεριλαμβανομένης μάλλον και της ε, προοπτικής, της ενδεχόμενης προοπτικής ε, διαμοιρασμού της ε, Συρίας σε διάφορες οντότητες, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο του διαμελισμού του Ιράκ αναφέρθηκε σαν ένα πολύ κακό σενάριο. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε το, επόμενο διάστημα. Επίσης να πω ότι παντού η ε, η συζήτηση ξεκίνησε ε, με αναφορά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ενώ ήξεραν ότι ερχόμαστε από την Ευρώπη, πάντα οι πρώτες συζητήσεις ε, ξεκινούσαν ε, για την νέα ε, διακυβέρνηση Τραμπ, για τα νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Τώρα βέβαια προέκυψαν, τα ξέρουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Από την πλευρά του Ισραήλ είδαμε μεγάλη αισιοδοξία είναι ευτυχείς γιατί βλέπουν ε, έναν φίλο του Ισραήλ και των Ισραηλινών. Εδώ να πω ότι ε, πολλοί ε, από τους Ισραηλινούς μας συνομιλητές μας κατηγόρησαν ότι έχουμε μια στάση ιδιαίτερος φίλο-παλαιστινιακή. Επίσης στη Ραμάλα βέβαια ακούσαμε πολλές ανησυχίες ε, και στο Αμάν ε, ε, κατά δεύτερο λόγο όσον αφορά τις θέσεις του Τραμπ ε, να σας ε, ε, θυμίσω ότι υπάρχει και μια σημαντική επίσκεψη του βασιλέως της Ιορδανίας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εκεί θα ξεκαθαριστούν ίσως περισσότερο κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει, η, θα αντιμετωπίσει ο Λευκός Οίκος την κατάσταση. Να σας πω ότι σε τρεις, στις τρεις μέρες ε, δεν έγινε καμία αναφορά στην αγαπητή Φεντερίκα Μογκερίνη. Ούτε μία φορά δεν ανέφεραν οι συνομιλητές μας το, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Κανένας δεν μίλησε ούτε για την κυρία Μογκερίνη, ούτε και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, λες και δεν υπήρχε. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ κυρία Πρέντα. Ο κύριος Παρσίνο. Παρνιό. Παρνιό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Παρνιό. Ε, μετά από αυτά που είπε ο πρόεδρος ε, ε, Μπρόκ και ο κύριος Πράντα, Πρέντα, συγγνώμη, δεν έχω πολλά πράγματα να πω, λέει ο κύριος Παρνιό. η λύση των δύο κρατών πραγματικά βρίσκεται σε κίνδυνο κυρίως στη Δυτική Όχθη, ε, το θέμα της, ε, του επικισμού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα πράγματα ε, περιπλέκονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, έτσι ώστε ο πολιτικός ορίζον που έχουμε και η λύση που θεωρούμε καλύτερη να απομακρύνεται όλο και περισσότερο ο Αγμέτ Τιμπή, τον οποίον μιλήσαμε, μας συζήτησε το θέμα και είπε ότι όσο ε, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις ε, των ε, Αράβων Ισραηλινών, τα πράγματα θα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο, θα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε λοιπόν για τα θέματα αυτά με τους συνομιλητές μας, μιλήσαμε με τον πρίγκιπα Φεϊζάλ της Ιορδανίας και εκείνος μας είπε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της, του μηνός Μαρτίου ε, θα συζητήσει το θέμα με, τους, ε, με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη. Ε, τώρα, όσον αφορά την κατάσταση, τη νέα κατάσταση με τον πρόεδρο Τραμπ, πραγματικά τα πράγματα περιπλέκονται και είναι δύσκολο να συνεχιστεί η, η, καταπολέμηση αυτή, αυτού του μίσους που διαπιστώνουμε. Κάτι άλλο το οποίο ε, μας ε, ε, έριξε τη σκιά του ας πούμε, ήταν το ψήφισμα 2334 ε, λίγες μέρες πριν και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να έχουμε και κάποιες ε, ε, συναντήσεις ε, οι οποίες θα ήταν στο ύψος της αντιπροσωπείας μας. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η σημασία της δράσης της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή το κενό το οποίο δημιουργείται μετά από την εκλογή Τραμπ θα πρέπει οπωσδήποτε να το καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το καλύψουμε εμείς. Θα πρέπει να προωθήσουμε και τα συμφέροντα όλων των λαών της ε, περιοχής ε, να ακουστεί η φωνή μας ε, γιατί η, εξωτερική, υπηρεσία εξωτερικής δράσης όπως είπε ο κύριος Πρέντα είναι απολύτως απούσα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τα πράγματα κύριε Πρόεδρε έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης σωστός ε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, επί του οποίου εργαζόμαστε μαζί με άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Καλά δεν είπα το όνομά σας, λέει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Απλώς να προσθέσω κάποια σημαντικά στοιχεία κατά τη δική μου την άποψη. Και εγώ συμφωνώ ότι η λύση των δύο κρατών δεν είναι πλέον βέβαιη. Δεν το βλέπω καν να πλησιάζει. Ήταν πολύ θλιβερή αυτή η επίσκεψη για μένα. Διότι συνειδητοποίησα και πάλι ότι η Παλαιστίνη, εντός του κράτους του Ισραήλ είναι ένας λαός που υποφέρει. Γιατί είναι δύο τα συστήματα που εφαρμόζει το Ισραήλ στην περίπτωσή τους. Ένα κράτος με δύο συστήματα. Ένα σύστημα για τους Ισραηλινούς και ένα δεύτερο για τους Παλαιστινίους. Να σας περιγράψω απλώς μία εικόνα. Ένα παράδειγμα στην Πιφλέμ. Μια εικονα ενα παραδειγμα στην τιφλεμ μια πολη με 180.000 κατοίκους, Παλαιστινίους, οι έπικοι του Ισραήλ, η Ισραηλινή έπικοι, είναι 100.000 μέσα στην πόλη την ίδια. Σαν ένας καρκίνος στο σώμα της πόλης. Και αρκετά με κομικό τρόπο δεν πληρώνουν καν το, το δημοτικό τέλη στο Δήμο της Βιθλέμ. Έχουν ένα δρόμο τον οποίο χρησιμοποιούν κάθε μέρα για να φύγουν από την περιοχή αυτή και εκεί δεν μπορούν καν να οδηγήσουν οι Παλαιστινοί, δεν έχουν το δικαίωμα. Δηλαδή πραγματικά μια χώρα με δύο συστήματα. Όποιο το λέει αυτό σε έκφραση, πραγματικά δεν περιγράφει την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό που προσπαθούσα εγώ δηλαδή να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται σαν μια δύναμη ήπια. Ίσως να είναι, αλλά όταν συμπεριφέρεται κανείς έτσι, ακόμη κι αν είναι ήπιος, ελαχιστοποιεί και μειώνει την ίδια της τη δύναμη. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει τον οποιονδήποτε ρόλο. Τον βασικό ρόλο πρώτα να αναλάβει ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μάλλον αυτόν τον, αυτός έχει τον βασικό ρόλο. Αυτός έχει την εξουσία και οι Παλαιστίνοι αναγκάζονται να αποστούν σοβαρότατη πίεση. Αυτό που βλέπουμε είναι για την ερχόμενη 20 ετία η κατάσταση να επιδεινώνεται δεν βλέπω να βρίσκεται λύση στην πράξη. Ακόμη και αν προσπαθήσει η Ρωσία, ακόμη κι αν ο κύριος Τραμπ πάει την πρεσβεία από, την, από το Τελαβή στην Ιερουσαλήμ, υπάρχουν τέτοιες φήμες, αλλά στην περίπτωση που κάνει κάτι τέτοιο, τα πράγματα θα επιδεινωθούν λίγο παραπάνω. Και βλέπουμε από την πλευρά των Παλαιστινίων να υπάρχει τάση ε, να επαναστατήσουν πάλι ε, και από την πλευρά των Αράβων. Εδώ λοιπόν νομίζω καλύτερο θα ήταν η κυρία Μογκερίνη να ήταν κάπως σαφέστερη. Πολύ περισσότερο σαφής και προς τις δύο πλευρές. Διότι υπάρχει πρόβλημα με τη ήλπιζα η Χαμάς και η Φατάχ να βρουν μια κοινή πορεία και όχι να λένε ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε γιατί είναι μία η εκπροσώπηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μέσεριτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπροκ και που διεύθυνε την διεξαγωγή της αντιπροσωπείας αυτής και για την πολύ καλή επισκόπηση που έκανε. Συμφωνώ με όσα είπατε και έχει περάσει η ώρα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σα τραβήξω περαιτέρω. Απλώ δύο πράγματα που θα θεωρώ σημαντικά για τη συνεδρίωσή μα εδώ, για τη συνεδρίαση, την κοινή συνάντηση στην ΚΝΕΣΕΔ. πραγματικά ήταν ευνηδιαστικό ότι στο σεμινάριο που είχε τίτλο η κατά δια την προσώπου πόλεμη μόνο η Ευρωπαϊκή Μάλλον στην, μόνο την ευρωπαϊκή πλευρά ακούστηκε αυτό. Από του άλλου δεν ακούστηκε καν η Σαουδική Αραβία. Σαν να ήταν ταμπού το όλο θέμα αυτό. Για μένα ήταν ε, κάπω ευνηδιαστικό. Και μετά μεσοπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε προοπτικέ. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο, αλλά το θέμα είναι ένα θέμα πραγματικά μα προκαλεί σύγκριση. Αν ρωτήσει κανεί τα μέλη τη Κινέσια, κυρίω από το κυβερνό κόμμα, εντάξει, ας πούμε ότι δεν δουλεύει η λύση των δύο κρατών. Τι άλλο πλάνο έχετε, τι εναλλακτικό πλάνο. Δηλαδή, ωραία, ας πούμε ότι η λύση είναι η λύση του ενός κράτους, αλλά θα πρέπει να είναι μια λύση δημοκρατική που να γίνονται σεβαστά τα ανθρωπινά δικαιώματα, όπως λέει ότι είναι το Ισραήλ, και να έχει και έναν ιουδαϊκό χαρακτήρα. Πώς αυτά τα τρία στοιχεία ταυτόχρονα θα περάσουν. Δεν έλαβα απάντηση. Μάλιστα σε μια από τις ε, άτυπες συνομιλίες που είχα, ε, μου δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αυτό που εννοούν με τη λύση του ενός κράτους είναι το status quo, το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Αυτό όμως δεν είναι βιώσιμο όπως ξέρουμε όλοι. Είναι ένας τρόπος να προκληθούν πάλι επεισόδια, να υπάρξει κλιμάκωση της βίας σε 5 ή 10 χρόνια. Και νομίζω πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να βρούμε ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ επί του θέματος. Διότι σε αυτή τη φάση απλώς κοιτάνε να κερδίσουν χρόνο για να διατηρηθεί το status κουβό. Δεν πιστεύω ότι θα διευκρινίσει το Ισραήλ από μόνο του πολύ σύντομα τη θέση του. Θα πάρει μήνε, για να μην πω ε, χρόνο, ε, για να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση Τραμπ επί του θέματο, αν δεν του πιέσουμε. Ευχαριστούμε και εμεί. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντε στι αντιπροσωπείε ήταν ο κύριος Ματουσχέλο, τουλάχιστον στο Ισραήλ, ο κύριος Αρνελίτς και ο κύριος Γιούρεκ απουσιάζουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω από πλευρά μου όλα αυτά που είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Για μένα το σημαντικότερο ήταν η τεράστια ανησυχία που ακούσαμε για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. Όχι μόνο για ε, ε, το κράτος του Ισραήλ, αλλά για ολόκληρο το αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ελμαρ Μπρόκ για την εξαιρετική του προεδρία και ήταν προνόμιο και τιμή για όλους μας να είμαστε μαζί του στην τελευταία αυτή αποστολή ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών. Ήταν συμβολικό που πήγαμε στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και στην Ιορδανία. Σε ευχαριστώ γι' αυτό, Έλμαρ. So. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την ενημέρωση για την συγκεκριμένη επίσκεψη. Πάμε στο 22 διάφορα. Όχι, προφανώς. 23. Προσεχή συνεδριάση 9 Φεβρουαρίου 2017, 9 η ώρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.